Διαβάζω την έκθεση της Επιτροπής για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταπολέμηση της απάτης. Εκεί τονίζουμε τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη για να ταυτίσουν και να καταπολεμήσουν τις ατασταλίες και απάτες καθώς και τις παρατυπίες που τουλάχιστον αυτές, τουλάχιστον αυτές που έχουν υποβληθεί στην Κομισιόν και περιπτώσεις υποψίας απάτης και κατάχρησης των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Για πρώτη φορά κάνουμε και συστάσεις πώς να βελτιωθεί η προστασία της χρήσης των χρημάτων του, Ευρωπαϊκού του Ευρωπαίου φορολογούμενου και φορολογούμενης. Η καταπολέμηση της απάτης και των παρατυπιών και ατασταλιών θεωρούμε ότι πρέπει να διασφαλιστεί, να συνοδευτεί από δύο άλλα επιτροπικά έγγραφα το ένα από αυτά παρουσιάζει τα στατιστικά στοιχεία σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια από ό,τι η συνθετική έκθεση. Η Κομισιόν εκτιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δημοσιεύει και δική του ετήσια, ε, δικό του ετήσιο ψήφισμα κατά των απατών. Πράγμα το οποίο έρχεται να συμπληρώσει την ετήσια έκθεση της Όλαφ η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη προσπάθησαν το συνολικό αποτέλεσμα των απατών αυτών όμως αυξήθηκε το 8 ήταν 1 δισεκατομμύριο 158 εκατομμύρια ενώ το 9 1.835 Όσο για τις υποψίες απατών και αυτές κατέληξαν σε πολύ περισσότερο, μεγαλύτερα ποσά. Ο ανατομέα δεν βρίσκουμε τις ίδιες τάσεις σε όλους. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση, ο αριθμός περιπτώσεων παρατυπίας στον τομέα των ιδίων πόρων και των αμέσων δαπανών έπεσε το 9 σε σύγκριση με το 8. Σε άλλους τομείς όπως η γεωργία, η πολιτική συνοχή και τα ταμεία προένταξης, τα προενταξιακά ταμεία, υπήρξε αύξηση στον αριθμό των παρατυπιών και των υποψιών απάτης. Αυτό εξηγείται από πολλούς παράγοντες μπορεί να δείχνει ότι τα συστήματα καταπολέμησης των απατών εργάζονται πιο αποτελεσματικά και γι' αυτό αναφέρονται περισσότερες περιπτώσεις. Θα αναρωτηθείτε βέβαια ποια είναι ακριβώς τα μέτρα που ελήφθησαν πέρυσι για να προστατευτούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Τα βασικά μέτρα που πήραν τα κράτη-μέλη το 9 τα βλέπετε στις προσθήκες της έκθεσης και συμπεριλαμβάνουν τροποποίηση της νομοθεσίας, της εθνικής νομοθεσίας για τις εθνικές προμήθειες, καλύτερη ανταλλαγή απόψεων και συνεννόηση των μεταξύ των αρχών, πιο αποτελεσματικές διαδικασίες επιστροφής χρημάτων, προγράμματα δράσης γενικά καταπολέμησης της απάτης. Εδώ επέμεινε ιδιαίτερα η Ουγγαρία, εκπαίδευση των τελωνιακών και άλλων δημοσίων υπαλλήλων και αυτά δεν είναι καν όλα. Έχω ήδη τονίσει από την αρχή ότι η Κομισιόν για πρώτη φορά έκανε συγκεκριμένες συστάσεις προς τα κράτη-μέλη στην, έκθεση, στην ετήσια έκθεση θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα τις εξής. Για την υποβολή παραπώνων ως προς τη χρήση του προϋπολογισμού πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νέο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του ίντερνετ για την υποβολή παραπώνων και πληροφοριών. Οι βελτιώσεις που απαιτούνται για τις επιστροφές και τους επιτοπίους ελέγχους, αυτές τις ανέφερα ήδη προηγουμένως. Πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή και σε θέματα όπως η έγκαιρη πληροφόρηση και υποβολή των στοιχείων και πληροφόρηση για τα μέτρα που ελήφθησαν. Την καταλληλότερη συνέχεια που θα δοθεί για τις συστάσεις αυτές θα τη δούμε σε λίγο, σε άλλα βήματα Ίσως να πρέπει να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό για την επιτήρηση και της εφαρμογής των συστάσεων αυτών. Πώς ακριβώς δηλαδή τα κράτη-μέλη θα λάβουν μέτρα για να προστατεύσουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν ίσως στην ετήσια έκθεση του 10. Θα τα δούμε όλα αυτά και στην επόμενη συνάντησή μας με την Όλαφ. Επίσης η Κομισιόν έχει εφαρμόσει και μόνη της, από μόνη της ορισμένα μέτρα αυτεπαγγέλτος όπως ένα πολιετές σχέδιο από το 9 και μετά για βελτίωση και των ε, ελέγχων. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών ΚΚΕ έχει ενδυναμώσει τη συνεργασία του με τρίτες χώρες και εθνικές οργανώσεις και διεθνείς οργανώσεις ιδιαίτερα με τον ΟΗΕ για να υπάρχουν πιο διαφανείς διαδικασίες. Η πρωτοβουλία αυτή επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών για τα προγράμματα που συγχρηματοδοτεί η Κομισιόν με τα κράτη-μέλη και τους διεθνείς οργανισμούς. Και τέλος θα ήθελα να αναφέρω ότι η Κομισιόν έκανε βελτιώσεις και στο δικό της σύστημα ελέγχου. Έχει ήδη προτείνει απλοποίηση των κανόνων λειτουργίας των διαρθρωτικών ταμείων και θα εξετάσει τη δυνατότητα και περαιτέρω απλοποιήσεων και σε άλλους τομείς. Η διεθνή συνεργασία ως προς την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και της καταπολέμησης των παρατυπιών, ατασταλιών και απατών έχει επίσης ενδυναμωθεί. Έχουν συναυθεί ορισμένες σημαντικές διεθνείς συμφωνίες ή πολυμερείς συμφωνίες που διαπραγματεύθηκε εκ μέρους της Ένωσης η Κομισιόν. Το 2009 η Επιτροπή Κομισιόν διαπραγματεύθηκε τις συνθήκες ένταξης της Ένωσης στην διάσκεψη για την καταπολέμηση των απατών διεθνώς που προτάθηκε από τον ΟΗΕ. Επίσης έχουμε υπάρξει πρωτοπόρος στην καταπολέμηση των διεθνών ε, φορολογικών παραδείσων. Ζητήσαμε από το Συμβούλιο εντολή για διαπραγμάτευση αναλόγων συμφωνιών και με την Ανδόρα, το Σαν Μαρίνο και την Ελβετία καθώς και το Μονακό. έχουμε διαπραγματευτεί με την Ουκρανία μια νέα συμφωνία στα πλαίσια της πολιτικής καλής γειτονίας για την καταπολέμηση της απάτης και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η διεθνής φορολογική συνεργασία με την Ουκρανία θα χρησιμοποιηθεί σαν βάση για τις μεραιτέρω διαπραγματεύσεις και με άλλες χώρες στα πλαίσια ε, συμφωνιών σύνδεσης και άλλων. θα προσβλέπουμε και στο μέλλον στη συνεργασία με σας και είμαστε έτοιμοι όπως και τα προηγούμενα χρόνια να συνεργαστούμε για προς το συμφέρον των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Ευχαριστώ. Κύριε Σεμέτα, θέλετε να μιλήσετε τώρα για το σημείο 15 της ημερήσιας διάταξης για την απαλλαγή 2009, τώρα ή μετά. Θα προτιμούσα να μιλάσουμε μετά τη συζήτηση του πρώτου κύριε Πρόεδρε. Α, με είχαν πληροφορήσει αλλιώ. Γι' αυτό σας ρώτησα. Δίνω το λόγο τώρα στον εισηγητή, στον κύριο Ιβαν. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, Επίτροπο για την υποβολή αυτής της έκθεσης. Όσον αφορά τις δαπάνες και τις ε, δημοσιονομικές επιπτώσεις που αναφέρατε, βλέπω να έχουμε μια, ένα διπλασιασμό το 2009 σε σχέση με το 2008. Αναφέρετε τα διάφορα στοιχεία. Το 2009 έχουμε πάνω από το 17 δισεκατομμύρια. Αναφερθήκατε στο θέμα της ε, πολιτικής συνοχής που έχουμε μια αύξηση της τάξης του 9%. Σημαντικά ποσά δηλαδή και σημαντικές αυξήσεις. Και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται με την εφαρμογή του συστήματος ε, διαχείρισης όταν υπάρχουν ατασταλίες. Ανακράτος μέλος και τομέα θα ήθελα να μου πείτε. Όταν συζητάμε τους ιδίους πόρους, αναφερθήκατε στην έκθεση για το 2010 και θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ σε αυτό. Πρόκειται για το προστευμένο τελευταίο σύστημα. Θεωρώ ότι θα ήταν καλό η Κομισιόν γλίγορα να εξετάσει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις των αποτελεσμάτων αυτής της έκθεσης και ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στους συμμετέχοντες οικονομικούς ε, παράγοντες που εργάζονται βάσει του απλουστευμένου αυτού συστήματος. Γιατί υπάρχουν πολλές ατασταλίες, περιπτώσεις μάλιστα απάτης που ανοιχνεύονται πολλές φορές μετά τις επίσημες προθεσμίες. Θα ήταν λοιπόν καλό να εξετάσουμε αυτό το σημείο, γιατί υπάρχει εδώ μεγάλος κίνδυνος. Και θα πρέπει οι υπεύθυνοι να κληθούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ταυτόχρονα θα ήθελα να αναφερθώ σε ασφαλείες για τους ίδιους σπόρους, όπου υπάρχει μία μείωση σχετικά με το 2008 στην έκθεση του περασμένου έτους το αναφέραμε αυτό όταν εξετάζαμε το θέμα της αποτελεσματικότητας των ελέγχων, ιδίω των ελέγχων για την παράνομη εισαγωγή ε, τηλεοράσεων. Επί θα ήθελα να αναφερθώ στην έκθεση του προηγουμένου έτους, όπου ζητήσαμε υπό αυτή. αυτοί Ε, να επανεισπραχθούν εφόσον έχουν χορηγηθεί βάση ατασταλιών. τα μία πραγματικά ανησυχητική η κατάσταση. Η Κομισιόν μόνο εν μέρη μπορεί να εξηγήσει τις τάσεις που παρατηρούνται. Για το 2006 είχαμε ε, ορισμένα αποτελέσματα. Τα σημερινά αποτελέσματα είναι ακόμα χειρότερα όμως. Αναφερθήκατε σε διάφορα στη... αριθμητικά στοιχεία όσον αφορά την ανάξη αυτών των αγριοστήρων καταβεβλημένων ποσών. Θα ήταν καλό ε, να μελετήσουμε τις πληροφορίες που δίνεται πολύ ωραία στην έξω του 2009, αλλά βλέπουμε ότι τα ποσοστά είναι πολύ ψηλότερα από το παρελθόν 44%. Υπάρχει λοιπόν πολύ δυνατότητα βελτίωσης. Και εν κατακλείδη, θα ήθελα να σας πω ότι εδώ έχουμε εν μέρη αύξηση των ασταλιών σε διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε και καλύτερη παρουσίαση, δηλαδή ε, οι αντασταλίες αυτές ανοιχνεύονται πολύ πιο καλά. Και θα ήταν λοιπόν καλό να μπορούμε να πούμε κατά πόσον αυτή η αύξηση των ασταλιών οφείλεται σε καλύτερη παρουσίαση και συλλογή των στοιχείων ή σε πραγματική αύξηση των ασθενειών. Σας ευχαριστώ. Αρχίζει η συζήτηση. Ο κύριος της πρώτος και καλύτερος. Κύριε Πρόεδρε, με κύριε Επίτροπε. Πραγματικά αυτές οι ατασταλίες, ιδίως στον τομέα της ε, πολιτικής συνοχής της Γεωργίας, και προναξιακό ταμείων και το θέμα της ανάκτησης αυτών των ποσών. Και αν διαβάσει κανένα την έκθεση του 2009, δημιουργείται η εντύπωση ότι εάν παραβλέψουμε την έκθεση 2007, θα χάσουμε την ευκαιρία να επανακτήσουμε κάποια δισεκατομμύρια ποσών που αγριοστήτως έχουν καταβληθεί. Χθε είχαμε τον διευθυντή της Όλαφ εδώ και δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι ορισμένοι ίσως ορισμένα σώματα δεν τολμούν να αναφέρουν τους λόγους για το οποίο υπάρχουν για οι αλλιές και γι' αυτό αυξάνονται. Ξότιμη κύριε Επίτροπε, καταλαβαίνω ότι ο τομέας των ευθυνών σας είναι πολύ ευρύς και ίσως έχετε και κάποιο όραμα για το τι θα μπορεί να γίνει στο μέλλον, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επανακτήσουμε αυτά τα ποσά που τους κατευρύθησαν. Ευχαριστώ κύριε Γκρέσλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον Επίτροπο για την έκθεση του αυτή που είναι πολύ εντυπωσιακή γιατί δείχνει πραγματικά και σημαντικές βελτιώσεις του συστήματος. Παραδείγματος χάρη το manager system που έχει ε, ανοίξει τώρα και που έχει βελτιώσει τον αριθμό των δηλώσεων παραδείγματος στον ερωτικό τομείο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν ε, τομείς ε, φαιοί και αριθμητικά στοιχεία που δεν βλέπουν το φως της ημέρας και πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε τα στοιχεία αυτά να τα ανοιχνεύσουμε. Η πρώτη μου ερώτηση είναι προβλέπετε κάτι τέτοιο και πότε. Δεύτερον, κάτι είπα και χθες τον κύριο Άιλετ. Είδα ότι η Γενική Γραμματεία που έχει προετοιμάσει την εκθεσία προσπαθεί να βρει τα ποσοστά απάτης. Θα ήθελα να ξέρω εσείς ως Επίτροπος πώς εκτιμάτε την αξιοπιστία αυτών των στοιχείων. Γιατί παραδείγματος χάρη βλέπω ότι για την Ιταλία υπάρχει 0,58, για άλλη μια χώρα 0,03. Αυτά τι νόημα έχουν. Είναι νομίζω σαν να λέμε ότι εντάξει δεν είναι και τόσο πολύ σοβαρό. Γιατί έχουμε τώρα και μία συζήτηση για το πόσο, είναι, πόσο υψηλός είναι ο ανεκτός κίνδυνος για τις απάτες. Ξέρω. Θεωριστικά συζητούμε το ένα και από την άλλη μια κάνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία υπόσταση. Έχω την εντύπωση δηλαδή ότι η έκθεση αυτή προσπαθεί να παρουσιάσει τα πράγματα λιγότερο σοβαρά από ό,τι είναι. Ε, τρίτη ερώτηση. Συμμετείχε η Όλαφ σε αυτή την έκθεση. Τέταρτη ερώτηση. Βλέπετε τα προβλήματα που υπάρχουν για την υπεραξή των αχρεωστήτων κατευθυνθέντων ποσών. Ε, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί όταν υπάρχουν αχρεωστήτως κατεβληθέντα ποσά, θα πρέπει τουλάχιστον να τα επιστρέφει κανένας. Και εάν είναι γνωστό ότι η πιθανότητα να επανεισπραχθούν τα ποσά, να επιστραφούν αυτά τα ποσά είναι πολύ χαμηλή, δηλαδή 20 με 30%, κανένας δεν φοβάται αυτό το μέσο. Θα πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε. Το έλαβα και υπόψη μου και στους ε, λογαριασμούς του 2009. Το καλοκαίρι αυτό ήταν ένα από τα κείμενα που μελέτησα και προσπάθησα να τα συγκρίνω με τα στοιχεία του Γενικού Διευθυντή για την περιφερειακή πολιτική, την αγροτική πολιτική ε, και με διάφορα άλλα έγγραφα και πάλι είδα ότι όσον αφορά το θέμα ποια χρήματα έχουν επιστραφεί στα διάφορα ταμεία, υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά στοιχεία εκάστοτε. Λοιπόν, οριστικά δεν ξέρουμε πόσα χρήματα πραγματικά επανακτούνται. Με το προκάτοχό σα ε, τον ε, και Επίτροπο το είχαμε συζητήσει, είχαμε ε, τσακωθεί για το θέμα αυτό, αν μπορώ να το πω έτσι. Υπάρχουν χώρες που 100% επέστρεφες. Λουξεμβούργο. Η Τσεχία όμως ε, κάτω από 8%, η δική σας χώρα κάτω του 5%. Στο κάτω-κάτω τμήμα βρίσκεται στην, ε, στον πίνακα αυτό. Τι γίνεται λοιπόν στην περίπτωση αυτή με, με τα κρατημέλη. Πέμπτη ερώτηση. Ε, τα κοινοτικά ταμεία πρέπει να προστατευτούν, αλλά πώς θα προστατευτούν τα εθνικά εκάστοτε ταμεία που χρησιμοποιούν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ας πούμε η βουλγαρική μαφία μας λέει ότι σταμάτησε τώρα να, να εξαπατεί με τα εθνικά χρήματα και περιορίζει τις απάτες στα εθνικά χρήματα, ε, μου φαίνεται ότι είναι κάπως περίεργα αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ο κύριος Σοντή, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την παρουσίαση και να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρόκειται για μια έκθεση για τις απάτες, αλλά μιλάμε πολύ στην έκθεση για τις παρατυπίες. Εγώ είχα πει παλιότερα ότι πρέπει να γίνεται μια διάκριση μεταξύ των απατών των και των λαθών όπως πρέπει να γίνεται και μεταξύ των απατών και των παρατυπίων, διότι στην απάτη υπάρχει η πρόθεση εμείς μπορούμε να, δεχόμαστε, να δεχθούμε μία διόρθωση ή μια παρατυπία δηλαδή δεν εφαρμόζουμε τον κανόνα ο κανόνας πολλές φορές είναι τόσο πολύπλοκος που οδηγεί στο λάθος, στην παρατυπία. Η απάτη όμως, για την απάτη πρέπει να έχουμε όμως την ανοχή μηδέν. Διότι ο πολίτης δεν μπορεί να δέχεται την απάτη. Ποια είναι η μάχη λοιπόν κατά της απάτης. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλές απάτες, στην έκθεση όμως κατανοούμε επίσης ότι υπάρχουν και πολλές παρατυπίες. Εγώ ως βουλευτής και πολίτης δεν, το αισθάνομαι εδώ ποια είναι η προβληματική για την απάτη και πώς την καταπολεμούμε. Επίσης μιλήσατε ε, κύριε Επίτροπε για τη σχέση με τη δικαιοσύνη. Χθες συζητήσαμε με την Όλαφ και είπαμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει απάτη, θα πρέπει να υπάρχει και προσφυγή στο ε, στη δικαιοσύνη, στο, στο ποινικό. Λοιπόν, πώς ε, τιμωρούνται οι απαταιώνες. Ευχαριστώ, δεν υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις, ο Επίτροπος. Σας κατευχαριστώ για τα σχόλια αυτά. Αρχίζω με το τελευταίο του κύριου Οντή. Πράγματι, είναι πολύ σημαντικό να διαχωρίσουμε την απάτη από μία απλή παρατυπία. Το επίπεδο απατών που ταύτισαν τα κράτη-μέλη είναι πολύ περιορισμένο. Κάτω του 1% ή και λιγότερο ακόμα των το συνολικών ποσών που κυκλοφορούν που χορηγούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία αλλά οι παρατυπίες βέβαια είναι πολύ περισσότερες και πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Μερικές ε, αφορούν απλώς ε, κακή χρήση, παραλήψεις εγγράφων, άλλες είναι πιο σοβαρές και πρέπει βέβαια να τα χειριστούμε όλα αυτά. Για το σύστημα διαχείρισης παρατυπιών εφαρμόζεται πλήρως στη γεωργία και αυτό μάλλον εξηγεί την αύξηση των παρατυπιών που έχουν ταυτιστεί στον τομέα αυτών γιατί το σύστημα επιτρέπει ακριβώς πολύ πιο αποτελεσματική υποβολή των παρατυπιών πληροφόρηση για αυτές. Έχουμε ζητήσει από όλες τις χώρες μέλη να εφαρμόσουν ένα παρόμοιο σύστημα και σε άλλους τομείς, σε όλους τους τομείς. Για τη συνοχή βέβαια είναι πολύ ψηλό το ποσοστό παρατυπιών και τρεις χώρες μέλη, η Γαλλία, η Ιρλανδία και η Ισπανία, δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει καθόλου το σύστημα. Σκοπεύω λοιπόν με τις υπηρεσίες μου βέβαια μαζί να συνεργαστώ με αυτά τα κράτη-μέλη που δεν έχουν εφαρμόσει το σύστημα και να τους ζητήσω να το πράξουν όσο το δυνατόν συντομότερα για να έχουμε καλύψει έτσι όλους τους τομείς που αφορούν την παρατυπία. για τις επιστροφές και τις χρηματικές διορθώσεις σύντομα ξέρω ότι θα συζητήσετε την έκθεσή μας για τους λογαριασμούς και μάλιστα για πρώτη φορά η Κομισιόν όπως σας είπα έκανε μια πολύ πιο λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης του τι συμβαίνει ως προς τις επιστροφές και έκανε και κατανομή ανακράτος Είναι πολλές οι πληροφορίες λοιπόν αυτές και επιτρέπουν την ανάλυση και την ανάληψη δράσης. Συμφωνώ απόλυτα ότι Η κατάσταση των επιστροφών σε επίπεδο κρατών μελών θα μπορούσε και θα έπρεπε να βελτιωθεί. Δεν έχω καμία αμφιβολία περί τούτου. Συνεχίσαμε τους επιτόπιους ελέγχους στα κράτη-μέλη και το θέμα της παρατυπίας ή μάλλον των επιστροφών, με συγχωρείτε λέει ο μιλητής, ήταν το κύριο θέμα των ελέγχων αυτών και σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη πέρασαν από αυτή τη διαδικασία και όσες δεν έχουν ακόμη περάσει θα το πράξουν φέτος μέχρι το Δεκέμβριο. Επίσης στην παρουσίασή μου σας είχα πει ότι υπάρχουν και πρόσθετες εγγυήσεις που θα έπρεπε να χορηγηθούν στα συμβόλαια όπως ε, καταθέσεις εγγυήσεων από τον ωφελούμενο ώστε να έχει και αυτός περισσότερη ευθύνη και να επιστρέφει τα ποσά εάν έχει αποδειχθεί κακή τους χρήση όσο δε για τον ενωσιακό προϋπολογισμό εμείς εφαρμόζουμε πολύ αυστηρά το σύστημα διορθώσεων ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα της Ένωσης. Συμφωνώ όμως ότι πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταλήγουμε στην επιστροφή όλων των χρημάτων που έχουν τύχει κατά Ακόμα το δουλεύουμε και θα το συνεχίσουμε. Η συνεργασία της Όλαφ στη σύνταξη της έκθεσης αυτής, η Όλαφ συνεργάστηκε και μάλιστα πλήρως έγραψε και δική της έκθεση και συντόνισε συντόνισε τις προσπάθειες των διαφόρων γενικών διευθύνσεων και άλλων υπηρεσιών. Δεν υπάρχει λοιπόν αφιβολία για τον ρόλο κλειδί που παίζει η Όλαφ και γι' αυτό. Αν δεν απατώμε αυτές είναι οι απαντήσεις που είχα να σας δώσω. Α, υπήρξε και το θέμα, θέθηκε το θέμα της συνοχής των παρατυπιών στον τομέα της συνοχής. Ναι. Πώς εξηγεί το υψηλός αριθμός παρατυπιών στη συνοχή. Το 2009 σημειώθηκαν τρεις περίοδοι, τρεις φάσεις παρατυπιών. 94-99 2000 με 2006 και 6 με 8. Για το 2000 με 2006 είμαστε στην τελευταία φάση της εξέτασης και οι έλεγχοι για παρατυπίες γίνονται ακόμα και έτσι εξηγείται η αύξηση του αριθμού των παρατυπιών. Γενικά όμως η κατάσταση στη συνοχή βελτιώθηκε πολύ σημαντικά κατά το 2009. Άλλος λόγος για τον υψηλό αριθμό παρατυπιών στη συνοχή είναι η Ρουμανία και η Βουλγαρία που μόλις άρχισαν να υποβάλουν στοιχεία για τις παρατυπίες των και είναι υψηλός ο αριθμός στις χώρες αυτές των παρατυπιών και αυξάνεται έτσι ο συνολικός αριθμός. Τώρα η παράληψη υποβολή στοιχείων, ναι. Εμείς περιγράφουμε την κατάσταση όπως φαίνεται από τα στοιχεία που μας δίνουν τα κράτη-μέλη και από δικές μας διαπιστώσεις. Δηλαδή διαπιστώνουμε κατά τις έρευνες της Όλαφ και τους ελέγχους από άλλες γενικές διευθύνσεις και εμείς στοιχεία παρουσιάζουμε δηλαδή τις πληροφορίες που διαθέτουμε όχι αυτές που δεν έχουμε δεν είμαστε 100% σίγουροι ότι έχουν υποβληθεί και γίνουν γνωστές όλες οι παρατυπίες που έχουν σημειωθεί και οι απάτες αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποκαλύψουμε στο Κοινοβούλιο όλες τις πληροφορίες που διαθέτουμε στη φάση αυτή. Αυτό εν συντομία, αυτά εν συντομία είναι αυτά που είχα να απαντήσω στις ερωτήσεις των αξιοτήμων κυρίων βουλευτών. Πάμε τώρα στο σημείο 15 της ημερήσιας διάταξης Απαλλαγή 2009, Γενικός προπολογισμό ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, Τμήμα 3 Επιτροπή και έχετε το λόγο για την εισαγωγή. Σύντομα βουλευτέ, κύριε και κύριοι, χαίρομαι που έχω τάση να σα παρουσιάσω ένα συμφαλεκτικό έγγραφο τη ε, διαχείριση του 2009 και την ετήσια έκθεση διαθέτηση για τους εσωτερικούς ελέγχους. Καταρχήν, η, τα επιτεύγματα στον τομέα της διαχείρισης ε, είναι ένα μέσο το οποίο αναλαμβάνει η Κομισιόν πολιτική ευθύνη και παρουσιάζει και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και τις ε, δράσεις που προβλέπουν για την βελτίωση της διαχείρισης και του γενικού ελέγχου. Αυτή η συνθετική έκθεση για το 2009 υιοθετήθηκε από τη νέα Κομισιόν. Αναλύει το έργο που έχει επιτεθεί από το 2009 για να προχωρήσουμε ε, και να παρουσιάσουμε τη δέσμευση των λόγων για το θέμα αυτό. Αναφέρεται εδώ το έργο για το 2009 σε διάφορα σημεία παραγωγής για τα τάσ μέσω των ε, εκθέσεων ετησιών δράσεων. Αναφέρονται επίσης ε, οι επιφυλάξεις που υπάρχουν. Σε γενικές γραμμές 20 επιφυλάξεις υπήρχαν στην έκθεση δράση του 2009 σε σχέση με 15 το 2008. 11 νέες επιφυλάξεις εκφράστηκαν το 2009 και 9 είχαν ε, συνεχιστεί από το περασμένο έτος. 9 από τις επιφυλάξεις, η, από τις 9 επιφυλάξεις η μία ήταν ε, για θέματα επανάληψης, το οι άλλες ήταν για ε, δημοσιονομική τέλεση. Έχουμε εδώ παραδείγματο χάρη το τομέα της έρευνας και το μη σεβασμό των κανόνων για τις δημόσιες αγορές και προμήθειες. Οι επιφυλάξεις οφείλονται σε, διάφορες, ε, ε, σε διάφορους λόγους, παραδείγματος χάνει καθυστέρηση στην εφαρμογή μεγάλων προγραμμάτων ε, πληροφορικής. Όλες αυτές οι επιφυλάξεις εξτάστηκαν από τι αρμόδιες υπηρεσίες και ελέγχθησαν και σε πρακτικό και σε πολιτικό επίπεδο. Η αύξηση του αριθμού των επιφυλάξεων είναι μια απόδειξη το ότι οι γενικοί διευθυντές γνωρίζουν σήμερα τις επιπτώσεις που έχουν στα, στον προπολογισμό όλες οι παρατυπίες, της αντισταλίσεις και απάτες. Μια περαιτέρω ένδειξη ότι οι αντιμετωπίζονται οι ρίζες των επιφυλάξεων είναι ότι η οικονομική έκθεση από τις επιφυλάξεις που μεταφέρθηκε από το 2008-2009 μειώθηκε κατόπιν της εφαρμογής των προγραμμάτων δράση υπό το φως των αποτελεσμάτων ε, ελέγχου του προπολογισμού μπορούσαν να έρθουν έξι επιφυλάξεις που αφορούσαν τη διαχείριση των ε, πόρων στη Βουλγαρία από το Γενικό Διευθυντή για την πολιτική διαβρύση και περιφερειακή πολιτική, η διαχείριση των πόρων στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία, ε, Γεωργία και Ράξης Πένθρου, Επίσης στον τομέα της ε, φυλακής πολιτικής και της αλληλείας τον έλεγχο του προγράμματος δαπανών για τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων. Ο κάθε φορά που έρετο μία επιφύλαξη, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης ε, παρουσίασε τις ε, πληροφορίες ότι το πρόγραμμα, πρόβλημα δηλαδή αντιμετωπίζεται επί τόπου. Στις περισσότερες περιπτώσεις είχε αυξηθεί σε επαρκές επίπεδο και το σύστημα ελέγχου ήταν το σωστό. Η Κομισιόν ε, αναγνωρίζει ότι χρειάζονται περαιτέρω βελτιώσει, ιδίω όσον αφορά για την ημερισμένη διαχείριση και στην κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών ε, χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαχείριση των κοινωτικών πόρων. Επίσης, ε, μέσα στα πλαίσια αναθεώρηση του δημοσιονομικού οικονομισμού, η Κομισιόν πρέπει να ελέγξει και να διευκρινίσει τις αρμοδιότητες κάθε φορέα και επίσης την δήλωση ασφάλειας που, σε του τομείς που δεν τεχάνουν τις άμεσες διαχείρισεις από την Κομισιόν. Αυτό θα βελτιώσει πολύ την εξασφάλιση των ε, ανησυχιών. Εγώ θα ήθελα να ενθαρρύσω τα κράτη-μέλη να αρχίσουν να κάνουν τις διάφορες δηλώσεις εξασφάλισης ε, ε, πριν προχωρήσει η αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Η Κομισιόν ε, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα όσον αφορά ιδίω τι δημόσιε προμηθειε που οδηγούν σε πολλέ πηγές σφαλμάτων έχει ήδη υποβάλει προβλήματα, ε, προτάσεις συγγνώμη, προσπαθώντας να μεταφερθεί σε ένα πιο απλό σύστημα, περισσότερη χρήση δηλαδή καταποκοπήν ποσών και καταποκοπήν ποσοστών. Επίσης υιοθετήσαμε μία ανακοίνωση με κάποιες φιλόδοξες προτάσεις για να απλουστευτεί η διαχείριση του τομέα της έρευνας. Λόγω των περιπλόκων κανόνων, η Κομισιόν ε, ε, πιστεύει θα πρέπει να εφαρμοστεί μια προσαρμογή ανοιχτού κινδύνου σφάλματος για να μην χρειαστεί να γίνουν περιττέρω ακόμα επενδύσεις στους ελέγχους. Θα ξαναέρθω στην Επιτροπή στις 15 Νοεμβρίου για να έχω μια εις βάθος ανταλλαγή μαζί σας ε, όσον αφορά το θέμα της ιδέας του ανοιχτού κινδύνου. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι δεν πρόκειται για ένα νέο κατόφλι βασιζόμενοι σε υγιείς εκτιμήσεις του κόστους των ελέγχων και εις βάθος έλεγχο των κινδύνων, η στρατηγική ελέγχου θα πρέπει να διαμορφωθεί αποτελεσματικά όσον αφορά το κόστος και όσον αφορά και το κίνδυνο. Να είναι απόλυτα σαφής κάθε φορά που υπάρχει ένα σφάλμα, θα πρέπει οπωσδήποτε αυτό να διορθώνεται, χωρίς εξέλιξη. Τον Μάιο του 2010 η Κομισιόν υπέβαλε την πρώτη της συγκεκριμένη πρόταση όσον αφορά το ελεγχόμενο επίπεδο κινδύνου για την έρευνα, την ανάπτυξη και τον ύπεθρο και την αγροτική ύπεθρο. Προσεχώ θα υποβάλλουμε για όλους τους τομείς συμπεριλαμβανομένους και τη συνοχή. Η Κομισιόν θεωρεί ότι όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να εξετάσουν τι προτάσει αυτέ. Ξέρουμε κύριε βουλευτέ, οι προσπάθειε που κατεβλήθηκαν τα πέντε τελευταία χρόνια για να βελτιωθεί η διαχείριση των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καρποφόρησαν. Βρήκαμε ποια είναι τα κύρια προβλήματα στη διαχείριση των Ταμείων και από την Κομισιόν και από τα κράτη-μέλη και υποβάλαμε συγκεκριμένε προτάσεις για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη βελτίωση. Χρειάζεται όμως και περαιτέρω δράση, όπως αναφέρθηκε στην ε, <coughs> ανακεφαλαιοτική αυτή έκθεση. Η Κομισιόν εστιάζει τις ε, προσπαθήσεις για να πετύχει αυτό που υπήρχε στις συστάσεις των ελεγκτών. Έχουμε τελικά εννέα επιτρόπους οι οποίοι ελέγχουν όλες τις ε, πολιτικές δαπανών. Αυξάνοντας την ε, γνώση του συλλογικού οργάνου της Κομισιόν των προβλημάτων αυτών, αυξάνει η Κομισιόν την πολιτική της ευθύνης αφορά τη διαχείριση του Προπολογισμού τη Ένωση από τι υπηρεσίε του. Επίσης, συμφωνήσαμε να εξετάσουμε περισσότερο την ε, ανάγκη μηδενικού ποσοστού κινδύνου. Επίση, ζήτησα από του εσωτερικού ελεκτέ να ελέγχουν σε όλε τι υπηρεσίε, όχι μόνο κατά πόσο έχουν εφαρμοστεί πλήρω τα προγράμματα δράση αλλά και κατά πόσον οι δράσεις που ενηλήφθησαν οδηγούν πραγματικά στην μείωση του κινδύνου. Πιστεύω ότι οι εσωτερικοί ελέγχοι θα πρέπει να συμβάλλουν ε, στο να βελτιωθεί η κατάσταση και να έχουμε θετικά DAS. Επίσης η Κομισιόν σημείωσε το αίτημα του ε, Κοινοβουλίου για την ανάγκη οργάνωσης ε, μιας διοργανικής διάσκεψης για το σύστημα απαλλαγής. Θα θέλαμε να οργανώσουμε αυτή την εκδήλωση το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους, ίσως τον Απρίλη. Θα ήθελα αυτό το, αυτή η εκδήλωση να χρησιμοποιηθεί για να ανοιχνεύσουμε πώς μπορούμε να βελτίσουμε την διαχείριση κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα αποτελέσματα των μελετών μας να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη μέσα στα πλαίσια και των προγραμμάτων για την οικονομική περίοδο που αρχίζει το 2013. Τώρα θα σας πω δύο λόγια για τις εσωτερικές ε, εσωτερικούς ελέγχους που έγιναν το 2009. Η έκθεση αυτή αφορά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι υπηρεσίες το 2009, τις συστάσεις που δόθηκαν και τις δάσεις που ενηλήφθησαν βάσει των συστάσεων αυτών. Συμπληρωμένα επίσης μη ένα κατάλογο των ε, τελικών ελέγχων από την ΕΑΕΣΤΕ τη στιγμή κατά την οποία ολοκληρώθηκαν αυτοί οι έλεγχοι. Η Κομισιόν ε, με ικανοποίηση σημειώνει ότι η αύξηση του ποσοστού των συστάσεων IS ε, είναι περίπου στο 99% και τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου όσον αφορά το αποτέλεσμα της IIS για την αντικειμενικότητα και τη συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας διαχείρισης και ελέγχου. Η Κομισιόν χαιρετίζει επίσης τη στρατηγική οργάνωση της ΑΕΑΕΣ σε στενή συνεργασία με τις δυνατότητες γενικών ελέγχων. Το 66% των δεσμεύεων του προπελισμού εμπλέκονται εδώ και το 100% των δεσμεύσεων για τους ελέγχους θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη του έτους. Οι κύριες συστάσεις του IIS για το 2009 αφορούν τη συνεχή της, ε, των επιχειρησιακών δράσεων και τη διαχείριση του κινδύνου, άμεσες ε, ε, χρηματοδοτήσεις, δημόσιες προμήθειες, εξωτερικές σχέσεις. Όσον αφορά τα μη δημοσιονομικά θέματα, η Κομισιόν αποφάσισε να μην δεχτεί πλήρω τι συστάσει που έκανε γενικό ελεγκτή όσον αφορά την ανάγκη αποκέντρωση ορισμένων ε, ελεγκτικών υποχρεώσεων. γιατί θεωρήσε ότι αν ανατεθούν οι ευθύνε αυτέ σε ένα κεντρικό σε μια κεντρική υπηρεσία θα μειωθεί η ευθύνη των γενικών διευθυντών. Ιδίω στο τομέα τη ε, πληροφορική, η Κομισιόν θεωρεί ότι έχει επιτευχθεί προοδρό σημαντική στου τομεί που ανείχνευσε η ΑΕΣ. Μία task force έχει οργανωθεί στο τομέα αυτό και εξετάζει τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Σε αφορά τα δημοσιονομικά θέματα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίε κομισιών έδωσαν τα κατάλληλα προγράμματα δράσης σαν αντίδραση στις συστάσεις που έχουν υποβληθεί. Ορισμένα από αυτά εφαρμόστηκαν ήδη, αλλά γενική εικόνα του επίπεδου εφαρμογής μπορεί να αξιολογηθεί μόνο με, τις, ε, ε, με τους επόμενους ελέγχους. Η Κομισιόν θα ήθελε να τονίσει ότι εξετάζεται ιδιαίτερα το θέμα αυτό όταν προσπαθούμε να βρούμε πώς θα μειώσουμε τις αδυναμίες και πώς θα βρούμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι όπως γίνεται μέσα στα πλαίσια της ανακεφαλικής έκθεσης. Τα προγράμματα δράσης θα πρέπει να είναι οργανωμένα στο επίπεδο κάθε γενικής διεύθυνσης. Αυτό ισχύει και για τη συνέχεια που δίνεται σε περιλαιότερες συστάσεις ΑΕΣ. που χρειάζονται πάνω από τους 6 μήνες για να εφαρμοστούν τις πιο σημαντικές δηλαδή. Η Κομισιόν θεωρεί ότι υπάρχει μια πολύ θετική εξέλιξη όσον αφορά το επίπεδο εφαρμογής. Παρ' αυτά πολύ σημαντικές συστάσεις ε, που έχουν καθυστερήσει πάνω από έξι μήνες καταδεικνύουν ότι υπάρχουν ακόμα καθυστερήσεις και αδυναμίες στην εφαρμογή των προγραμμάτων δράσης. Η Επιτροπή ε, των Ελέγχων κατηγορία ότι δεν έχουν ληφθεί αρκετά μέτρα για να εφαρμοστούν αυτές οι παλές συστάσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και μπορώ ευχαριστώ να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Τώρα ο λογιστής της ε, Κομισιόν, ο κύριος Μπράιαν Γκρέι, ο ελεγκτής λογιστής της Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έγινε η παρουσίαση της θεσμικής μας έκθεσης που βασίζεται στα συγκεκριμένα δεδομένα που σας στείλαμε όπως είμαστε υποχρεωμένοι. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα βασικά. Απλώς αν έχετε ερωτήσεις να απαντήσω. Ευχαριστούμε. Ο εισηγητής κύριος Χατζημαρκάκης. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Σμέτα και τον κύριο Γκρέι για τις παρουσιάσεις τους αυτές. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε κάτι, γιατί ακριβώς η αδυναμία των ε, εκθέσεων αυτών είναι ότι είναι εκθέσεις κάθε γενικής διεύθυνσης. Ε, το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε, ε, όπως το παρελθόν στην Επιτροπή, μέχρι την Επιτροπή Σαντέρα, που υπήρχε μια γενική παρουσίαση, ένα γενικός έλεγχος. Τώρα έχουμε εκθέσει κάθε μιας γενικής διεύθυνσης που βέβαια είναι, δεν είναι από ανεξάρτητο ελεγκτή που κεντρικά προετοιμάζει αυτές τις εκθέσεις. Η κάθε γενική διεύθυνση υποβάλλει τις εκθέσεις και εσείς ε, μετά κάνετε αυτή την ε, εγκεφαλοκητική έκθεση. Το θέμα είναι ποιος ελέγχει τους γενικούς διευθυντές. Γιατί από εκεί και πέρα η υπογραφή του γενικού διευθυντή ε, επιβεβαιώνεται αν θέλετε με μια υπογραφή του συλλογικού οργάνου απλώς. Δηλαδή έχουμε κατά κάποιο τρόπο οργανωμένη ανευθυνότητα γιατί κανένας επίτροπος δεν ελέγχει ο ίδιος τον γενικό του διευθυντή. Θα ήθελα να μου το εξηγήσετε αυτό γιατί έχω την εντύπωση ότι πραγματικά από την Επιτροπή πρώτη και εδώ βρισκομε, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία εκμάθησης, όπως φαίνεται και από την ε, συγκεφαλαιολογική σας έκθεση, που στην σελίδα 5, στο αγγλικό κείμενο, υπάρχει έτσι ένα, μια δήλωση που λέει ότι η Κομισιόν θα συνεχίσει να εργάζεται για τη βελτίωση των ετησίων ε, ε, τον ε του περιοχικού μέσου με το οποίο οι κύριοι διατάκτε λογοδοτούν στο σώμα και ω πηγή αποδεικτικών στοιχείων για την ΕΕΔ. Κάλεσε επίση τη Γενική Γραμματεία και την Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού να εξακολουθούσαν να δίνουν κατευθυντήριε οδηγίε στι γενικέ διευθύνσει και στι υπηρεσίε, για τεχνική επανεξέταση των πάγιων εντολών, των καυτηρίων οδηγιών, των προγραμμάτων επιμόρφωση των συνεδριάσεων επανεξέταση ή από ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο κρίνουν χρήσιμο. Τέλο, καλωσού γενικού διευθυντέ και του προσταμένου τη υπηρεσία να υποστηρίξουν δραστήρια όλα τα μέτρα που λαμβάνουν οι κεντρικέ υπηρεσίε για να βελτιώσουν την ποιότητα των ΕΕΔ. Ετησίων εκθέσεων δραστηριοτήτων. Αυτό στη σλίδα 6 του κειμένου ε, καταδεικνύει ότι Καταβάλλω προσπάθειες για βελτίωση. Αλλά από όσο ξέρω, η Κομισιόν τις προσπάθειες αυτές καταλαμβάνει εδώ και πολλά χρόνια. Το ότι ακόμα βρισκόμαστε σε μια διαδικασία βελτίωσης με εκπλήτη. Θα έπρεπε να έχετε προχωρήσει κατά εδώ μου πολύ περισσότερο. Και έτσι τίθεται και διάφορα ερωτήματα καταρχήν γιατί η μέθοδος ελέγχου που εφαρμόζετε εσείς διαφέρει τόσο πολύ από τη μέθοδο ελέγχου του Ελεκτρικού συνεδρίου. Σύντομη απάντηση παρακαλώ και την θέμα αρχής. Δεύτερον, η επιφυλάξη, ο οποία ε, αναφέρθηκε και ο Επίτροπος μετά, που μας είπε το 2008 μέχρι το 2009, υπήρχε μια αύξηση επιφυλάξεων από το 15 στο 20. Λοιπόν, το 2008 είχαμε 15 μόνο από πληρώσεις γενικών διευθύνων Τώρα έχουμε 20 επιφυλάξεις. Αυτό καταδεικνύει αφενός ότι λαμβάνεται υπόψη πολύ σοβαρά η εσωτερική έλεγχη. Καλό αυτό. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν κατάλαβα ακριβώς πότε άρεται αυτές τις επιφυλάξεις. Τι κάνει η Κομισιόν, πού είναι το κατόφλι στην έκθεσή σας λέτε ότι έρονται αυτές οι επιφυλάξεις όταν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση. Τι θα πει επαρκής. γιατί ξέρουμε ότι θα κάνουμε τη συζήτηση για τον ανοιχτό κίνδυνο και ξέρουμε ότι η Κομισιό αυξάνει το επίπεδο αυτό και αναρωτιέμαι αυτό το επαρκώς ε, ικανός και λοιπά πώς το ερμηνεύεται. Πότε άρεται μια επιφύλαξη, γιατί ίσως αυτό αμφισβητήσει και όλη την έκθεση. Από ποιο κατόφλι και μετά θα αμφισβητήσετε όλη την έκθεση μιας γενικής γραμματείας. Επίσης, έχω και μια λεπτή ερώτηση να υποβάλω, που πρόκειται στις μεγάλες ε, χώρες μέλη. Είπατε κύριε Επίτροπε, ότι βρισκόσαστε σε μια συνεχή διαδικασία ενθάρρυνσης των κρατών μελών για καλύτερη συνεργασία. Και το Κοινοβούλιο οπωσδήποτε είναι εγγυητής ότι θα σας βοηθήσει. Θα με ενδιαφέρει όμως πόσο μεγάλη είναι η επίδραση μεγάλων κρατών μελών εσωτερικά και όταν γίνονται οι έλεγχοι. Σε περίπτωση που υπάρχουν διακυβεύονται σημαντικά κονδύλια, Παραδείγματο σαν Γαλλία και γεωργικό τομέα. Θα με ενδιαφέρε κατά πόσον ο αρμόδιο γενικό διευθυντή στον αγροτικό τομέα που είναι Γάλλος κάνει πραγματικά με τον ίδιο ζήλο τους ελέγχους αυτού στη Γαλλία όπως σε άλλες χώρες κατά πόσον εξετάζεται λεπτομερώς το θέμα αυτό, γιατί εμείς έχουμε κάποια μηνύματα ότι ασκείται πίεση από τις μεγάλες χώρες μέλη να μην είναι τόσο σοβαρή αυτή η έλεγχη. Σας παρακαλώ, μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Έχοντας εξετάσει προσεκτικά τις επιφυλάξεις, βλέπουμε ότι σε μεγάλους τομείς δαπανών υπάρχουν θέματα τα οποία συνεχίζονται πολλά χρόνια, παραδείγματος χάρη Άγιαξ και Ελλάδα πολλά πολλά χρόνια. Το 2009 έχουμε κάτι το καινούριο, που για μένα είναι πολύ αξιόλογο. Δηλαδή από τις δαπάνες για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Βλέπουμε τώρα να υπάρχει μια μετατροπή στον ουρατικό τομέα, δηλαδή εγκαταλείπουμε την μεμονωμένη ε, υποστηρίξη και υποστηρίζουμε την ε, χρηματοδότηση για την ίδια την υπαίθρο. Και εδώ δεν παίζει τόσο ρόλο η Άζαξ ε, όπως προηγουμένως. Και αναρωτιέμαι τώρα, θα αλλάξετε και τις μεθόδους ε, ελέγχου. Θα πρέπει να συζητήσετε βέβαια και με τον συνάδελφο Τόλος. Αναρωτιέμαι κατά πόσον η Κομισιόν θα πρέπει να ασχολείται με αυτό τον σημαντικό τομέα. Τι θα κάνει εδώ και άμα βρίσκεται σε διαδικασία επιμόρφωσης θα ήθελα να σας πω ότι εμείς ως Κοινοβούλιο θα εξετάσουμε τα θέματα πάρα πολύ προσεκτικά. Και μία ερώτηση προς τον κύριο Γκρέι. Συμφωνείτε ότι δεν υπάρχει κανένας κεντρικός έλεγχο, τελικός έλεγχος των εκθέσεων των γενικών διευθυντών και γι' αυτό δεν υπάρχει και κανένας που να αναλαμβάνει την ευθύνη. Κατά τη γνώμη, μας, τη γνώμη σας, συγγνώμη, ποιος θα ήταν ένα πιο αποτελεσματικό όργανο ελέγχου. Γιατί τελικά δεν υπογράφει ο Επίτροπος σε μετά, αλλά το συλλογικό όργανο. Και γι' αυτό μπορούμε να συζητάμε για οργανωμένη ανευθυνότητα. Παρόλε τι επικρίσει αυτέ, χαίρομαι πάρα πολύ για την συνεργασία μαζί σα όσον αφορά την απαλλαγή 2001. Ο κύριος Σίβεν. Ε. Εγώ θα είμαι σύντομο. Κι εγώ. Ο κύριος Χατζημαρκάκης μας έκανε την έκθεσή του για το πράγμα για το οποίο τον ευχαριστώ, αλλά υπάρχουν ορισμένα προβλήματα. Είμαι ικανοποιημένος από όσα έκανε για τη διαχείριση η Κομισιόν το 9, αλλά δεν μπορώ να πω το ίδιο και για τη διαχείριση των χωρών μελών. Και γι' αυτό υπάρχουν πολλοί λόγοι. Καταρχάς, μιλάμε για πολλές αλλαγές ως προς τα κριτήρια εκλογιμότητος. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ασχολούμαστε με πολύ πολύπλοκη μεθοδολογία. Και οι αλλαγές αυτές δεν ήταν και οριστικές, διότι όλοι ξέρετε ότι πρόκειται σύντομα να εφαρμοστούν νέες άλλες αλλαγές. Αυτό ισχύει και σε ενωσιακό επίπεδο και σε κρατικό. Η απλοποίηση των κανόνων και η περισσότερη διαφάνεια θα ήταν κάτι πολύ θετικό για να μπορέσουν οι εθνικές αρχές να διαχειριστούν τα ταμεία καλύτερα και αυτό θα βοηθήσει και τους ε, όσους ωφελούνται από αυτά γνωρίζουμε ότι ένας δημόσιος υπάλληλος που διαχειρίζεται εθνικά ευρωπαϊκά ταμεία είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει πάρα πολλούς κανόνες και γι' αυτό σημειώνονται οι καθυστερήσεις. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ αργή και μακρόσυρτη και γι' αυτό αναπόφευκτα καταλήγουμε και σε παρατυπίες και λάθη. Υπάρχει και άλλο πρόβλημα όμως που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, δηλαδή το πρόβλημα των δημοσίων προμηθειών. Και εδώ ισχύουν ιδιαίτερα πολύπλοκοι κανόνες. Ταυτόχρονα όμως οι κανόνες αυτοί αφορούν και εξαιρέσεις. Και αυτό είναι πρόσθετο βάρος, γιατί και αυτές αλλάζουν πάρα πολύ συχνά και οι αλλαγές γίνονται και από την Κομισιόν και από τα κράτη-μέλη. Στη Ρουμανία τα κριτήρια εκλογιμότητος ας πούμε άλλαξαν τη στιγμή που εγκρινόταν τα σχέδια. Και χρειάζονται όλο και νέα κριτήρια να προστίθενται και πολλοί αποκλείονται αδικαιολόγητα από τα κριτήρια. Πρέπει εδώ η Κομισιόν να είναι πιο αυστηρή έναντι των εθνικών αρχών, διότι η αλλαγή των κανόνων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ωφελεί ορισμένους και αποκλείει άλλους. Μερικές φορές η διαδικασία αυτή είναι πολιτική, γνωρίζουμε εκ των προτέρων δηλαδή ποιος θα ωφεληθεί από τη διαδικασία. Τέτοια πράγματα πρέπει να σταματήσουν. Θέλω να μου πείτε αν έχετε πληροφορίες για την εξέλιξη των πραγμάτων ως προς την διόρθωση προβλημάτων για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία για τις επιστροφές. Ποια είναι η θέση της Κομισιόν ως προς αυτό. Υπάρχουν κυρώσεις ή όχι. Ευχαριστούμε κυρία Γκρέσλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας πω ότι καμιά φορά έχω και εγώ αυτή την εντύπωση του Δηλαδή διαβάζω σε εκθέσεις αυτές, νομίζω ότι τα έχω ξαναδεί και τα έχω ξαναδιαβάσει. Δύο ερωτήσει. Όσον αφορά το IAS. Το ένα αφορά το Schengen, το όργανο Schengen. Και θα ήθελα να ξέρω πού βρισκόμαστε με αυτό. Ήταν και τμήμα τη τελευταία απαλλαγή το ε, κοινοβούλιο είχε κάποιες απαιτήσεις σχετικά προς το ελεκτικό συνέδριο. Στο έγγραφο εργασία Κομισιόν βλέπουμε τώρα μια, ένα σκιαγράφημα από την ε, δραστηριότητα του Γενικού Διευθυντή του 2008. Ότι υπάρχει περασμένη διαχείριση, εντάξει, αλλά όπως παρουσίασε αυτή τη στιγμή δεν μας ικανοποιεί και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γκρέι τι θα γίνει τώρα τελικά. Πότε θα εξαφανιστεί αυτό το θέμα πια από την ουσία μας διάταξη γιατί θα έχει επιληθεί. Η Κομισιόν κάνει ό,τι πρέπει χωρίς να κρύβεται πίσω από την πλάτη των κρατών μελών. Επίσης το θέμα του Άμπακ όπου ήταν τότε υπεύθυνο ο κύριο Γκρέι. Ε, μήπως υπάρχει εδώ μια σύγκρουση φερόντων τι έχετε να πείτε από αυτό. Ευχαριστώ ο Επίτροπος, ο κύριος Σεμέτα για τι απαντήσει. Σα ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και τι παρατηρήσει. Καταρχήν τονίζω ότι εδώ συζητάμε δύο εκθέσεις, δύο. Η μία είναι έκθεση δημοσιονομικού ελέγχου γενικότερα και η δεύτερη είναι σύνθεση των ετησίων δραστηριοτήτων και εκθέσεων από το Γενικό Διευθυντή, από τη Γενική Διεύθυνση. Στην συνθετική αυτή έκθεση παρουσιάζουμε μία σύνοψη, σύνθεση των ετησίων εκθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης και αυτό αποτελεί το κύριο εργαλείο του λογιστηρίου. Για να υπογραφεί δηλαδή πρέπει ο κάθε γενικός διευθυντής να λάβει υπόψη του όλες τις πηγές πληροφοριών της υπηρεσίας του και τους δημοσιονομικούς ελέγχους που έχουν γίνει και από την εσωτερική υπηρεσία της Κομισιόν. Όλες τις διαπιστώσεις πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό την ευθύνη αυτή να την έχει η Γενική Διεύθυνση, διότι πριν από μερικά χρόνια το πρόβλημα ήταν στην Κομισιόν ότι κανείς δεν ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση. Ενώ τώρα μπορούμε να ταυτίσουμε την ευθύνη του Γενικού Διευθυντή κάποιας συγκεκριμένης γενικής διεύθυνσης. Αυτό είναι σημαντική πρόοδος. Και αυτό θα συνεχιστεί και θα ενδυναμωθεί αυτού του είδους η διαχείριση, δηλαδή η υπεύθυνη διαχείριση. ο εσωτερικός διορθωσιονομικός ελεγκτής της Κομισιόν κάνει ελέγχους στις γενικές διευθύνσεις και γενικότερους παρατηρεί και κάνει συστάσεις προς τις γενικές διευθύνσεις που είναι υποχρεωμένες να λάβουν υπόψη τους. Ίσως ο Μπράιαν Γκρέι μπορεί να προσθέσει τίποτα επ' αυτού. Για την άρση των αμφιβολιών είναι κάτι πολύ σημαντικό και αυτό στη διαχείριση, στο διαχειριστικό σύστημα σύμφωνα με το οποίο αν μια γενική διεύθυνση εκφράσει αμφιβολίες πρέπει ο διευθυντής αμέσως να υποβάλει και ένα σχέδιο δράσης για του πώς προτίθεται να διορθώσει τα προβλήματα που ταύτισε. Στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων του. Είναι αποκλειστικά ευθύνη της κάθε γενικής διεύθυνσης να κρατήσει ή να άρει τις αμφιβολίες που έχει εκφράσει αλλά είναι υποχρεωμένος επίσης να κρίνει, να αποτιμήσει και πώς θα διορθώσει το πρόβλημα. Πρέπει να δει δηλαδή και ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους εκφράζει αμφιβολία ή για τους οποίους έρει την αμφιβολία αυτή. Για την επιρροή και σημασία των κρατών μελών. Και οι μεγάλες και οι μικρές χώρες μέλη, τουλάχιστον αυτές που αναφέρατε, προσπαθούν να κάνουν καλύτερη διαχείριση των ενωσιακών ταμείων. Και οι καθαροί εισφορείς ιδίω ενδιαφέρονται πάρα πολύ τα ενωσιακά χρήματα να χρησιμοποιούνται και να τυχαίνουν σωστής διαχείρισης. Προφανώς λοιπόν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα και η βελτίωση της διαχείρισης. άλλα θέματα απλοποίησης ότι μάλλον δηλαδή δεν αρκεί η απλοποίηση που έχει ήδη γίνει είπατε. Υποβάλαμε τις προτάσεις της απλοποίησης για τον τομέα της συνοχής, για την έρευνα και Κάναμε σειρά προτάσεων για απλοποίηση και στους δημοσιονομικούς κανονισμούς και συμφωνώ απόλυτα ότι όσο απλούστεροι είναι οι κανόνες τόσο πιο εύκολο είναι για τους χρήστες να ωφεληθούν από τα κριτήρια εκλογιμότητας. Αργότερα φέτος θα κάνουμε και μια ανακοίνωση για περαιτέρω απλοποιήσεις με βάση τις αναλύσεις και τις διαπιστώσεις μας για να δούμε τι άλλο θα μπορούσε να απλοποιηθεί στην προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περίοδου. Είναι σημαντικό εκ των προτέρων να δούμε ποιοι κανόνες θα μπορούσαν να απλοποιηθούν για την επόμενη περίοδο. Για τις δημόσιες προμήθειες και τους κανόνες τους συμφωνώ ότι είναι πολύ πολύπλοκο το σύστημα και οι κανόνες και θα έπρεπε και εδώ να βρούμε λύσεις για απλοποίηση. Ελπίζω να ακουστούν προτάσεις και στην ανακοίνωση που σας ανέφερα. Για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία είχαμε αμφιβολίες ως προς τη λειτουργία του έαντος του Άγιαξ και ζητήσαμε να μας πούν συγκεκριμένα πώς μπορούν να βελτιώσουν τα πράγματα και η Βουλγαρία-Ρουμανία έκαναν προτάσεις. Η Γενική Διεύθυνση ΓΕΟΡ διαπίστωσε πάντως σοβαρές παραλήψεις στην εφαρμογή του ΕΑΝΤΟΣ στη Βουλγαρία και Ρουμανία. Για το Σέγγεν, σύστημα πληροφόρησης Σέγγεν. Αυτό είναι γνωστό πρόβλημα και παλαιό. Δυστυχώς δεν λειτουργεί ακόμη πολύ καλά. Τι έκανε λοιπόν η Κομισιόν, ερωτηματικό. Βελτίωσε την πρόσβαση και τις δομές όπως τη δια, ηλεκτρονική διαχείριση των δεδομένων από τον χρήστη και σε για τις περιπτώσεις καθυστέρησης πρόβλεψε πρόστιμα. Πρόστιμα. Δεν μπορώ βέβαια να σας εγγυηθώ ότι έχει λυθεί το πρόβλημα των καθυστερήσεων, αλλά οι τελευταίες δοκιμές που κάναμε για τη σταθερότητα του συστήματος ήταν θετικές και από ό,τι ξέρουμε το σύστημα θα εφαρμοστεί. Και τώρα δίνω το λόγο στον Brian Gray. Σας ευχαριστώ, Επίτροπε. Το κύριο ερώτημα είναι η διακυβέρνηση της Κομισιόν και το θέμα του κεντρικού ελέγχου. Η ευθύνη των εσωτερικών ελεγκτών σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους πρότυπα επίσης είναι να ελέγξουν γενικά το θέμα της κυβέρνησης του οργάνου που εξετάζουν, τη Κομισιόν στην προκειμένη περίπτωση. Και εξετάζουμε κατά πόσον είναι πραγματικά υπεύθυνοι γενικοί διευθυντές για αυτό που κάνουν. Και αυτές οι Συλλογικέ εκθέσεις αντικατοπτρίζονται στην έκθεση του Γενικού Διευθυντή τελικά και υποβάλλονται στην Κομισιόν. Εκστάζουμε τη διαδικασία αυτή. Το 2006 είχαμε κάποια σχόλια. Ο Γενικός Γραμματέας και οι άλλοι άμεσα ενδιαφερόμενοι συμφώνησαν να ε, εισαγάγουν προγράμματα τράση για να βελτιώσουν τη μέθοδο με την οποία προετοιμάζονται οι ε, κεφαλαιοτικές εκθέσεις ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο τα, το όργανο συλλέγει τις εκθέσεις αυτές των ε, γενικών διευθυντών ε, και πώς τα υποβάλλει κλπ. ήταν τελικά ικανοποιητική. Εμάς, εμείς κοιτάζουμε και τι υπογράφουν οι επιμέρους γενικοί διευθυντές. Όλα αυτά τα στοιχεία για διακυβέρνηση είναι βάσιμα. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να υποβάλει τα στοιχεία που έχει στα χέρια του. Γιατί αισθάνεται τόσο σίγουρος για τα στοιχεία που υποβάλλει στο συλλογικό όργανο. Αυτό το κάνει λόγω της ε, δυνατότητας που έχει για εσωτερικούς ελέγχους. Και επίσης όσον αφορά την ε, οδηγία για τους σπόρους που πρέπει να υπογραφεί επίσης. Δηλαδή ο Γενικός Διευθυντής έχει την γενική ευθύνη, αλλά υπάρχουν μέσα οι γενικές ευθύνσεις και άλλοι οι οποίοι έχουν κάποιες δυνατότητες. Όταν λέμε βελτιώθηκε η διαδικασία, έχω να σας πω ότι αυτό που κοιτάει η ΑΕΣ είναι κατά πόσο αυτές οι εκθέσεις είναι σωστά ε, οργανωμένες, κατά πόσο μειώνουν το κίνδυνο και κατά πόσο βελτιώνουν καλύτερα πραγματικά τη διαχείριση του προπολογισμού. Εξετάζουμε επίσης τον τρόπο με τον οποίο ε, δημιουργείται η συγκεφαλαιοτική αυτή έκθεση. Δεν είναι απλώς μια προς... Ε, ένα άρθισμα των 41 εκθέσεων, αλλά για κάθε γενική διεύθυνση καθόμαστε γύρω από το τραπέζι και με τους γενικούς διευθυντές και εμείς ε, και εξετάζουμε ποια είναι τα προβλήματα που είχαν και ποιες είναι οι επιφυλάξεις που εκφράζουν. Αυτή η διαδικασία δηλαδή υπάρχει για, την, ε, για το έλεγχο της ποιότητας. Όταν καλύπτει το συλλογικό όργανο να εγκρίνει την ε, ε ανακεφαλωτική έκθεση υπάρχει μια διαδικασία που προηγείται που η ΑΕΣ ε, έχει εγκρίνει τις εκθέσεις αυτές. Βέβαια θέλουμε να μειώσουμε τις ευθύνες που έχουν ε, στις γενικές διευθύνσεις. Και γι' αυτό ε, η δική μας έκθεση που σας παρουσίασε από τον κύριο Σεμετά παρουσιάζει ορισμένους από τους κινδύνους που ενέχεται αυτή, αυτού του τύπου η διακυβέρνηση και τονίζουν ιδίως αυτήν την έκθεση του 2009 το τι θα πρέπει να γίνει όσον αφορά την ε, διαχείριση διαχείριση, τη συνέχιση τη διαχείρισης θα γίνει αν υπάρχει πια σφωτιά το περλεμό ας πούμε. Και λέμε ότι χρειάζεται βελτιωμένο συντονισμός κατά βάση σε κεντρικό επίπεδο. Το κεντρικό επίπεδο θα πρέπει να φροντίσει κάθε γενική διεύθυνση να γνωρίζει τι θα πρέπει να γίνει χωρίς να κάνει τη δουλειά ε, των γενικών διευθύνσεων το ίδιο. Έχουμε το θέμα της πληροφορικής παραδείγματος. Αν κάθε γενική διεύθυνση έχει το δικό της ε, σύστημα, <clears throat> δεν είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει και το εξαρτάζουμε με τη βοήθεια των, ε, των ερευνών που κάνουμε. Και η Γενική Διεύθυνση του, του Γενικού Γραμματέα έχει έναν δικό προπελισμό για να βελτιώσει την κατάσταση. Βέβαια, βελτιώνουμε, έχουμε βελτιώσει, πάντα μπορούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω. Και όπως είπε, είπε, όπως είπε ο ίδιος ο Επίτροπος, το 99% των συστάσεων βασίζονται σε αξιόπιστα προγράμματα. Όσον αφορά τα θέματα που έθιξε η Δόκτωρ Γκρέσλε για το Σέγκεν, είδαμε ότι η αρμόδια γενική διάθεση είχε εργαστεί πάρα πολύ καλά γιατί κατέγραψε τα προβλήματα στην Βουλγαρία και στην Ρουμανία και εξέτασε γιατί. Επειδή υπήρχε καθυστερημένη εφαρμογή, αργή εφαρμογή. Γιατί θα έπρεπε να δημιουργηθούν τα απαραίτητα ε, κυβερνητικά και δεσμικά όργανα, τόσο ώστε οι χώρες αυτές να δαπανούν τα χρήματα αξιόπιστα. Και η αρμόδια γενική διεύθυνση ε, έδρασε λογικά. Για το ΆΜΑΚ ε, γνωρίζετε, έχετε δίκιο. Η Άζαξ. Ε, ε, καλό είναι νομίζω. Καλό είναι το σύστημα αυτό. Υπάρχουν δύο πτυχές βέβαια. Το ένα είναι ο, η έλεγχη που επιβάλλει και εγώ συνέλεξα με τους συναδέλφους μου για να δω κατά πόσον αυτοί έλεγχοι εφαρμόζονται σωστά από τις άλλες υπηρεσίες, αλλά όσον αφορά το σύστημα ελέγχων αυτό καθ' αυτό, δεν ασχολήθηκα εγώ με τους ελέγχους, οι συνάδελφοί μου το έκανε αυτό χωρίς εμένα και το υπέβαλαν στην Επιτροπή Προόδου των Ελέγχων χωρίς να έχω συμμετάσχει εγώ καθόλου. Λοιπόν, μετά από ένα χρόνο νομίζω δεν υπάρχει πια σύγκρουση συμφερόντων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χατζημαρκάκη ζήτησε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και τον κύριο Γκρέμι για τα τόσο σωστά που μας είπαν εδώ. Ε, πιστεύω ότι υπάρχει ένας μηχανισμός, το αναγνωρίζω. Το να αποκολλείτε εσείς έναν υγιή μηχανισμό. Εγώ θα έλεγα ότι είναι καλά λαδωμένος αν θέλετε. Λειτουργεί πολύ καλά, αλλά κατά πόσο είναι ο ιδανικός μηχανισμός δεν ξέρω, γιατί είπατε ακριβώς ότι αυτή η έλεγχη είναι εσωτερική, εσωτερική στη γενική διεύθυνση. Και είναι σαφές, το ξέρουμε, όταν ε, παραδείγματος χάρη υπάρχουν εξετάσει σε μία τάξη ας πούμε, ε, υπάρχει εσωτερική διαδικασία. Είναι όλοι φιλικοί δηλαδή προς τη δική τους γενική διεύθυνση. Ε, είναι διαφορετική κατάσταση αν υπάρχει ένα εξωτερικός έλεγχο που γίνεται έτσι και από το ελεκτικό συνέδριο. Δεν θέλω να σας κατηγορήσω ότι υπάρχει κάποια επίδραση από αυτού, αλλά ψυχολογικά διαφέρει αν ο έλεγχος γίνεται από τους ίδιους συναδέλφους. Μετά είπατε, καθώς καθόμαστε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πραγματική κεντρική η μέθοδος ελέγχου όμως. Και είπατε ότι λίγα θέματα υπάρχουν τα οποία ε, καλύπτουν περισσότερες της μιας γενικής διευθύνσης, όπως το παραδείγμα χάρη η πληροφορική. Εμείς στην Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσουμε τι γίνεται. Χαίρομαι που ε, εκθέτει το θέμα τόσο ανοιχτά, γιατί ο κύριος Σιωμετά δεν ήταν έτσι κι αλλιώ υπεύθυνο για το μηχανισμό αυτό. Τον βρήκε, πρέπει όμως να συμμορφωθεί. Και γι' αυτό θα ήταν καλό από κοινού να προσπαθήσουμε να δούμε ποια είναι τα ποσοστά το σε ένα εσωτερικό σύστημα ελέγχου. Σα ευχαριστώ όμω για τη συνεργασία σα. Είναι πολύ καλή η βάση συνεργασία που μα προτείνετε. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τέμπους Φούγκιτ, παρακαλώ σύντομα. Ευχαριστώ πρόεδρε για την υπομονή σας. Άκουγα τον κύριο Χατζημαρκάκη και φαίνεται ότι δεν θεωρεί πολύ σημαντικό τον κοινοβουλευτικό έλεγχο του Κοινοβουλίου. Διότι οποιαδήποτε εταιρεία θα ήταν θα έκανε αυστηρότερο έλεγχο από τον εξωτερικό δημοσιονομικό που κάναμε εμείς. Ιδίως τώρα μπροστά σε αυτή την κρίση. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε και τους εξωτερικούς και τους εσωτερικούς ελέγχους. Πρέπει να πληρούν τα κριτήρια. Ωραία. Σας ευχαριστούμε. Επίτροπε Σιμέτα και κύριε Γκρέι και τώρα περνάμε στο σημείο 17 του κυρίου Σκυλακάκη ο οποίος όμως ζήτησε αναβολή για το τέλος της πρωινής συνεδρίασης Πάμε λοιπόν στο 18. Χορήγηση εγγύηση ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη μειών από δάνεια και εγγυήσει για σχέδια εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 18 ο λόγο έχει ο εισηγητή κύριο Θωμά Ντόιτ. Είπαμε αναβλήθηκε και το 16 είχε αναβληθεί. Δεν το θυμάστε, είχε αναβληθεί ήδη λοιπόν ο κύριο Θωμάς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδελφέ, το σχέδιο γνωμοδότησης που έχετε μπροστά σας αφορά τις εξωτερικές δραστηριότητε Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων από δάνεια και για σχέδια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις ζημίες που μπορεί να έχουν απορρεύσει από αυτά. Αυτό είναι το θέμα της νομοδότησης. Και έχουμε και τις τροπολογίες μου που συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο. Θα γνωρίζετε ίσως ότι ότι οι εγγυήσει του προϋπολογισμού προς την ΕΤΕ διασφαλίζουν τη σταθερότητα της τράπεζας αυτής και καλύπτουν τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι χώρες από τις δραστηριότητες της τράπεζας αυτής, ιδιαίτερα χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε δάνεια από τις αγορές. Υπάρχει κάποιο όριο κάποιο ανώτατο όριο για τη χρηματοδότηση που χορηγείται από την ΕΤΕ, 25,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Και οι χώρες που επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσουν είναι σε ένα γνωστό κατάλογο. Στις τρέχουσες δημοσιονομικές προοπτικές και κατά τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρησή τους αποφασίστηκε να δοθεί μια νέα εντολή που να καλύπτει όλες τις χρηματοδοτήσεις μεταξύ 2007 και 2013 και τα νέα στοιχεία της εντολής είναι τα εξής. 2 δισεκατομμύρια ε, προαιρετική εντολή για την καταπολέμηση των αποτελεσμάτων των κλιματολογικών αλλαγών και οι προηγούμενοι στόχοι θα αντικατασταθούν από καινούριου οριζόντιους στόχους. Υποδομές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλες βελτιώσεις. Η Κομισιόν σε διαβούλευση με την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων θα συγγράψει κατευθυντήριες γραμμές για κάθε περιφέρεια Επίσης θέλουμε να ενδυναμωθεί η δυνατότητα η δυνατότητα των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών στόχων και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε θέματα υγειονομικά, περιβάλλοντος, διαχείρισης υδάτων, αποχέτευσης, περιορισμού των αποτελεσμάτων κλιματικών αλλαγών κλπ. Τέλος, Θέλουμε να ενεργοποιηθεί η εξωτερική εντολή της ΕΤΕ για την Ισλανδία, τη Λευκορωσία και την, Καμ... την Καμπότζη και τη Λιβύη. Οι τροπολογίες σκοπεύουν ακριβώς την ενδυνάμωση των λειτουργιών ελέγχου του προϋπολογισμού με τρεις προτεραιότητες. Μεγαλύτερη διαφάνεια όλες οι εκθέσεις δηλαδή που αφορούν τις δραστηριότητες της ΕΤΕΝ να προωθούνται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεύτερον, τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Εγγυήσεων να, ή μάλλον που διαθέτουν Ευρωπαϊκή Εγγυήση να συνοδεύονται από μία έκθεση των αποτελεσμάτων τους. Και, και να είναι γνωστό και ποιος μπορεί να ελέγξει. Τώρα υπάρχουν πέντε τροπολογίες, πέντε τροπολογίες για τις τρεις προτεραιότητες, όπως προείπα. Για να δούμε λοιπόν τι λένε. Τι είδατε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και για τη συνεργασία με το προσωπικό της Επιτροπής και τη ΕΤΕ. Ευχαριστούμε. Κανένα σχόλιο ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, α, εντάξει, τότε περνάμε στην ειδική ευρωπαϊκή έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και αποτίμηση του αντικτύπου στα θεσμικά όργανα, ο εισηγητής κύριος Όλμπριχτ. Κυρίες και κύριοι, στο έγγραφο εργασίας μας, μου μάλλον, αναφέρομαι Συνειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αξιολογήσεις αντικτύπου στα δεσμικά όργανα της ΕΕ στηρίζουν τη λήψη αποφάσεων ερωτηματικό». Η έκθεση λοιπόν αυτή αφορά την ανάλυση του αντικτύπου όπως λέει και ο τίτλος και τους τρόπους χρήσης αυτού του εργαλείου, πώς εφαρμόζεται και τα λοιπά. Θέλω να τονίσω ότι στην έκθεσή του το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τονίζει ότι οι νομοθετικές προτάσεις της Κομισιόν συνοδεύονται από αξιολογήσεις αντικουτύπου, Αλλά και όμως Αυτές οι αξιολογήσεις αφορούν τις υποβληθήσεις προτάσεις. και άρα μετά γίνονται τροπολογίες, συζητήσεις και από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και αποτέλεσμα είναι το τροποποιημένο κείμενο να μην γίνεται αντικείμενο αξιολόγησης αντικού Αυτή είναι η διαφορά. Το συνέδριο επίσης λέει στην έκθεσή του ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κάνουν δικές τους αξιολογήσεις αντικτύπου. Δικές τους. Αλλά τα στοιχεία που έχει το συνέδριο λένε ότι αυτό έχει γίνει πολύ λίγες φορές σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Άρα βασικά οι αξιολογήσει αντικτύπου είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο το οποίο όμως δεν χρησιμοποιείται και τόσο συχνά, μπορεί και καθόλου. Μόνο στην πρώτη φάση της νομοθετικής διαδικασίας. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ιδιαίτερα τις συστάσεις της έκθεσης του συνεδρίου. Η Επιτροπή μας θα ήθελα να εγκρίνει τις συστάσεις αυτές. Πρώτα πρώτα λοιπόν, οι νέες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη νέων διαθεσμικών συμφωνιών. Όπως αυτού θα έπρεπε να ξανασκεφτούμε το εύρος και την ανάλυση των αξιολογήσεων αυτών αντικτύπου. Το αναφέρει η ισχύουσα διαθεσμική συμφωνία, αλλά στην πράξη φαίνεται ότι χρειάζονται αλλαγές του μόντους οπεράντη μας. Και εγώ το υποστηρίζω αυτό, το υποστηρίζω. Διότι οι αξιολογήσεις αντικτύπου πρέπει να συνοδεύουν νομοθετήματα και την νομοθετική διαδικασία σε όλες τις, τις φάσεις. Όποτε λοιπόν η Κομισιόν υποβάλλει κάποια πρόταση πρέπει πριν κατατεθούν οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να υπάρχουν και αξιολογήσεις για να ξέρουμε ποιοι ακριβώς είναι οι κίνδυνοι και οι αντίκτυποι των τροπολογιών αυτών. Βασικά δηλαδή, εδώ μιλάω για για πολλαπλές αξιολογήσεις. Πολλαπλές. Που πρέπει να κατατίθενται πάντοτε με την ίδια μέθοδο και να μπορούμε εκ των υστέρων να βλέπουμε ποιες είναι οι αλλαγές που προτείνονται. Πρέπει να έχουμε συνέστηση για τις επιπτώσεις των τροπολογιών που εμείς προτείνουμε. Αναρωτιόμαστε επίσης αν αυτή η μελέτη επιπτώσεων θα πρέπει να γίνεται από την Κομισιόν ή αν θα πρέπει το Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με αυτό. Αν εμείς επιλέγαμε τη δεύτερη λύση, το Κοινοβούλιο θα, μελέ θα ζητούσε μελέτη επιπτώσεων με διαφορετική μέθοδο από αυτή της Κομισιόν. Η πρόταση λοιπόν θέλει η Κομισιόν να κάνει την μελέτη επιπτώσεων μετά την κατάθεση των τροπολογιών. Επίσης, είναι ουσιαστικό να αυξήσουμε τη διαφάνεια, δηλαδή πρέπει να δημοσιεύονται τα αποτελέσματα των, της μελέτης επιπτώσεων, πρέπει να υπάρχει ε, ευρία πρόσβαση στην ε, μελέτη της αξιολόγησης των επιπτώσεων. Θα πρέπει επίσης να προβλέπονται πολλές δράσεις, κυρίως όταν πρόκειται για νέες νομοθετικές πράξεις που αφορούν είτε στην επιτροπολογία είτε στην απολούστευση. Είναι θεμελιώδες όλες αυτές οι προτάσεις να ακολουθούνται από μία μελέτη επιπτώσεων. Στο έγγραφο εργασίας που αναφέρεται και στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, εγώ ως εισηγητής προσπαθώ να καταστήσω κατανοητό ότι η αξιολόγηση των επιπτώσεων, η παρουσίαση δηλαδή των συνεπειών της κάθε πρότασης πρέπει να είναι μια σταθερή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίως μετά από τη θέση σε ισχύ της Λισαβόνας. Θα πρέπει να βλέπουμε λοιπόν, θα πρέπει μάλλον να διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για ένα πλέον έκτημα όχι μόνο για τον εισηγητή για την και για την πρόταση, αλλά και για όλο το κοινοβούλιο. Αυτό είναι το έγγραφό μου, σας το παρουσιάζω και οι εκπρόσωποι του ελεκτικού συνεδρίου μπορούν να, να το λάβουν υπόψη. ο κύριος Ενρίκ Κετά. Η Κομισιόν έχει θέσει ένα σε, σε ισχύ ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανάλυσης επιπτώσεων και λαμβάνεται υπόψη συνολικά από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα Μπορούν όμως να γίνουν βελτιώσεις όσον αφορά στις βασικές διαδικασίες, το περιεχόμενο και την παρουσίαση των εκθέσεων όπως το υπογράμμισε και ο εισηγητής σας. Το ελεκτικό συνέδριο ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα να παρουσιάσουν αυτήν την πρόταση κυρίως όταν έχουν κοινές νομοθετικές πράξεις των οποίων πρέπει να αναλύουν τις επιπτώσεις. Η κυρία Τσέσκοβα. Σας κατευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την πρωτοβουλία. Μέσα σε ένα μόλις χρόνο που είμαι εδώ στο Κοινοβούλιο συνάντησα, αντιμετώπισα τόσο πολλές φορές το πρόβλημα οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κομισιόν να βασίζονται σε καλές προθέσεις αλλά αργότερα να διαπιστώνεται ότι οι πρωτοβουλίες αυτές είναι διαστρεβλωμένες, διαστρεβλώνονται, αλλάζουν και χάνεται η αρχική πρόθεση. Πάρα πολλές φορές το έχω δει αυτό και ελάχιστες κατάφερε η Κομισιόν να πετύχει αυτό που πρότεινε πράγματι. Προφανώς το θέμα δεν λύγει σήμερα, αλλά πάντως το σημαντικό είναι να υποστηρίξουμε την πρόταση αυτή. Γιατί πιστεύω ότι όντως αυτές οι αξιολογήσεις αντικτύπου πρέπει να γίνονται με την ίδια μεθοδολογία. Ευχαριστώ. Thank Γιάννης Βάτσον. Uh, θα ήθελα να πω ότι και εμείς δεχόμαστε με μεγάλη χαρά την έκθεση του συνεδρίου που είναι πολύ χρήσιμη για μας και για τα τρία θεσμικά όργανα, όχι μόνο για την Κομισιόν αλλά και για το Κενοβούλιο και το Συνεβούλιο. Οι διαπιστώσεις του είναι πολύ χρήσιμες ως προς το πώς νομοθετούμε και παίρνουμε πολύ σοβαρά την πρότασή τους για βελτιώσεις. Μάλιστα πολλές από τις συστάσεις αυτές ήδη τις έχουμε συμπεριλάβει στον τρόπο εργασίας μας, στη μεθοδολογία μας. Κάτι που φαίνεται σαφέστερα από την έκθεση αυτή από ό,τι από προηγούμενες είναι ο ρόλος του Συμβουλίου και Κενοβουλίου. Και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε ακόμη περισσότερο τους επόμενους μήνες για την Κομισιόν υπάρχει η ανησυχία υπάρχει μάλλον η κοινή ευθύνη να κάνουμε την αξιολόγηση του τι σημαίνουν τα νομοθετήματα του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου ως προς την λειτουργία ας πούμε των επιχειρήσεων. Τώρα το πώς ακριβώς γίνεται η αξιολόγηση των αντικτύπων ενό νομοθετήματος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε προσεκτικά. Υπάρχει η διαθεσμική ισορροπία που καθορίζεται από τις συνθήκες και που καθορίζει σαφώς το ρόλο του κάθε οργάνου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν ώστε κάθε μας απόφαση να μην αντιτίθεται στην πρόθεση του νομοθετήματος και οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου πρέπει να προσέχει η Κομισιόν ποιες αντικτύπους έχουν. Να το παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας αυτό ως προς την τελική μας απόφαση. Πάντοτε λέγαμε ότι είμαστε έτοιμοι να σας πούμε ποια είναι η μεθοδολογία μας και επίσης έχουμε προσφέρει, προσφερθεί πολλές φορές να κάνουμε πρόσθετες αξιολογήσεις αν το ζητήσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεν το ζήτησαν πολλές φορές αλλά σε αυτή τη βάση μπορούμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Γενικότερα πάντως ως προς το πώς θα οργανώνουμε τις αξιολογήσεις στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αυτό είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε πολύ προσεκτικά τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε η κυρία Γκόλτμαγερ. Έχω μία πρόσθετη ερώτηση για την Κομισιόν. Είστε διατεθειμένοι γενικότερα να παίρνετε τα έγγραφα και να κάνετε την αξιολόγηση κάθε φορά αλλά να το γνωστοποιείτε και στους κοινοβουλευτικούς γιατί θα μας ήταν πολύ χρήσιμο γιατί έτσι έτσι μόνο μπορούμε να γνωρίζουμε ποια είναι η άποψη της Κομισιόν που είναι πάντα διαφορετική από των χωρών μελών, ιδίως ως προς το κόστος. Είναι τόσο διαφορετική που πολλές φορές με έχει εκνευρίσει. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε τα έγγραφα αυτά, παρακαλώ. Γενικά μπορείτε. Μάλιστα μπορούν να διατίθενται και αυτόματα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Συχνά λοιπόν πολλές φορές είναι ε, εμπορικά ευαίσθητες αυτές τις πληροφορίες και υπάρχει απόρριτο αλλά γενικά Αυτές οι πληροφορίες διατίθενται, μπορούν να διατεθούν και έχετε κάθε δικαίωμα να τις δείτε, να τις ζητήσετε. Παρόλα αυτά εδώ θίξατε ένα σημαντικό πρόβλημα της αξιολόγησης όχι μόνο του κόστους αλλά και του ωφέλους των νομοθετημάτων και εδώ πρέπει ακόμη να γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος. Εμείς το ξέρουμε πάντως, έχουμε συνείδηση και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιωθεί η ποιότητα των ποσοτικών μας στοιχείων. Γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχουν και όρια στο τι μπορούμε να κάνουμε στην Κομισιόν. Διότι εδώ βλέπουμε έχουμε 27 χώρες μέλη που πολλές φορές έχουν τεράστιες διαφορές και ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσουν μια νομοθεσία όχι μόνο ως προς το κόστος, αλλά και ως προς τις επιπτώσεις στην κοινωνία τους. Εδώ υπάρχει μια άλλη διαπίστωση του συνεδρίου ότι τα, ε, οι αξιολογήσεις που κάνουν τα κράτη-μέλη επίσης μπορούν να είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μέχρι τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μόνη χώρα που το κάνει αλλά είναι κάτι που και άλλες χώρες μέλη θα μπορούσαν ε, εποφελώς να κάνουν και να πληροφορούν βέβαια στο Συμβούλιο για τη θέση τους και ίσως και στο Κοινοβούλιο. Γιατί εξορισμού έχουν στενότερη σχέση με τους ενδιαφερόμενους για το θέμα του κόστους μιας νομοθεσίας και άρα μπορούν ευκολότερα να κάνουν και την ανάλυση. Είναι και αυτό μια σύσταση του συνεδρίου με την οποία συμφωνούμε απόλυτα. Να κάνουν τα κράτη-μέλη με καλύτερη προσπάθεια και τα ίδια να πληροφορούν πανενοσιακώς για τους αντικτύπους. διπλωματικότατη απάντηση αυτή της Κομισιόν αλλά αφού μιλάμε για πιθανές λύσεις, εδώ απαιτείται νέα διαθεσμική συμφωνία. Διότι ένα από τα συμπεράσματα είναι πώς θα γίνονται οι αξιολογήσεις μετά την τροπολόγηση μιας πρότασης. Μετά την τροπολόγηση πριν την έγκριση. Πολύ δύσκολο και διότι δυναμικό. Απαιτούνται λοιπόν νέες στάσεις και είναι εδώ και ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων που είναι και αυτός καινούριο με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας. Μπορούν και αυτά να αντιδράσουν μέσα στη διαδικασία. Πριν δείξουμε λοιπόν την κίτρινη κάρτα, για να το πω έτσι, πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση, δηλαδή οι προτάσεις να συμφωνούν με, την, με τον καινούργιο τρόπο λειτουργίας των θεσμικών οργάνων. Απαιτείται συμφωνία μεταξύ όλων των οργάνων και ένα από τα συμπεράσματα του συνεδρίου είναι ότι πρέπει όλα αυτά να είναι γραμμένα και με εύληπτο και ευνόητο τρόπο για να μπορούν να τα διαβάσουν και όλοι και όλες. Όχι μόνο οι αξιολογήσεις της Κομισιόν να γράφονται και να διαβάζονται από την Κομισιόν αλλά και από όλους και όλες τους πολίτες και τις πολίτησες. Το καλή για την επίσκεψη στην Ελλάδα. Δυστυχώ οι Έλληνε συνάδελφοι αυτή τη στιγμή αποουσιάζουν. Μια που όμω γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση στην Ελλάδα, θέλω να σα πω ότι η επίσκεψη ήταν πάρα πολύ σημαντική. Αυτά που είδαμε ήταν πάρα πολύ λυπηρά. Το είπατε και εσεί τώρα, κύριε Πρόεδρε, ότι οι απαντήσει τη νέα κυβέρνηση ε, δεν ήταν σαφεί. Ήταν πολύ λυπηρά αυτά που έγιναν επί σειρά ετών και θα πρέπει νομίζω να αναφερθεί αυτό ξεκάθαρα. Δεν βοηθάει τους Έλληνες εάν εμείς ε, τα παραβλέπουμε αυτά και διπλωματικά λέμε εντάξει θα περάσουμε στη... στο παρασύνθημα. Ακριβώς στον τομέα ΕΡΑΚΣ το είδαμε αυτό. Ήταν ένα θέμα όπου η Ελλάδα πολλά χρόνια ανήθηκε να εφαρμόσει ό,τι έπρεπε να εφαρμόσει και υπέκυψε μόνο στην πίεση της δικής μας Επιτροπής. Το λέω ξεκάθαρα, η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα που υποφέρει από την διαφθορά. Υπάρχουν και άλλες. Αλλά η Ελλάδα οπωσδήποτε είναι μια χώρα που έντονα και λόγω τη κρίση που ζει ε, πλήττεται ιδιαίτερα από την διαφθορά. Ο Πρωθυπουργό ε, Παπανδρέου το παραδέχτηκε όλο. Φαίνεται αυτό και στην έκθεσή μα. Και θεωρώ αν το παραδέχεται αυτό ξεκάθαρα η μια χώρα ότι υπάρχει συστηματική διαφθορά, θα πρέπει να αποφασίσουμε να το πούμε ξεκάθαρα. Δεν επιτρέπει να συγχύσουμε έτσι. Και απογοητεύτηκα και όπως μας αντιμετώπισε ο πολιτικός κόσμος που δεν μας έδωσε ξεκάθαρες αποφάσεις. Ένας συνάδελφος, ο κ. Σκυλακάκης, που δεν μπορούσε να ήταν εδώ, απεκλήφθη από το κόμμα του περασμένη εβδομάδα, είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, απεκλείστη λέω γιατί είναι υπέρ του μεταρρυθμιστικού προγράμματος που προωθούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ταμείο και το ε, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καταλαβαίνετε, απεκλείστηκε επειδή ήταν υπέρ. Λοιπόν, εμείς καλούμεθα τώρα να το πούμε αυτό ξεκάθαρα. Ενώ θα συνεχίσουν τα πράγματα όσοι έχουν η Ελλάδα τρία χρόνια θα μπορέσει να επιστρέψει τα χρήματα αυτά. Συνεχίζεται ε, να υπάρχει αυτή, αυτή η υπόσχεση, αλλά τελικά δεν θα γίνει τίποτα. Βλέπω εκεί την, ε, της, ε, ε της, αλλά δεν έχουν χρήσει πάρα πολύ, γιατί ίσως είναι οι ίδιοι εκείνοι που δρούνε ένα άλλο κόμμα, ίσως, αλλά είναι τα ίδια κόμματα που ε, διοικούν και αλλάσουν ε, τις, ε, τις μεθόδους, δεν τις αλλάσουν δηλαδή επαρκώς. Λοιπόν, έχουμε ένα τεράστιο σχέδιο, το ευρώ, και θα ήθελα να παρακαλώ στους αδέρφους να απαρνηθούν την διπλωματία και να πούν στους Ελληνές σκληρή αλήθεια για να τους βοηθήσουν. Αλλιώς δεν θα βοηθήσουμε ούτε εκείνους ούτε εμάς. Ευχαριστώ. Μια που θέλουμε να λέμε τα σιγά σιγά και σκάφη σκάφη, είμαστε διπλωμάτε εμεί. ήταν επιτυχη η επισκεψή μα γιατί είπαμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Εγώ θα ήθελα ότι έγινε ο τέος ε, διευθυντή από εκεί που ήταν υπεύθυνο για, την, για το κοινοβούλιο τότε και είχε δοθεί κάποιε υποσχέσει στου υιοργού ότι δεν θα χρειάζεται πια να υποβάλουν αιτήσει ε, ε, επίσημα όταν εκλεγεί. Αυτό είναι τελείως αντίθετο με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δεν μπορεί να μοιράζει τα χρήματα έτσι σε όποιον του αρέσει. Δεν θέλω να ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Ο γενικός ε, διευθυντής για την Γεωργία δεν είχε θέση εκεί επιφύλαξη, αλλά θέλω να το ξέρω αυτό. Λοιπόν, εδώ εκείνοι που είναι από την Κομισιόν εδώ θα ήθελα να το καταγράψουν αυτό και να το έχουν υπόψη τους στο αργότερο στη συνάντηση με τον Επίτροπο Τσόλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. για αρκετό χρόνο, πετυχαίνουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Χωρίς όμως την άσκηση της πίεσης αυτής, δεν θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Νομίζω αυτό είναι ένα θετικό αποτέλεσμα από την Ελλάδα για τη δική μας εργασία. Όσον αφορά τα νέα κράτη-μέλη, εγώ είχα προβλήματα με την έκθεση του Γενικού Διευθυντή Γεωργίας. Την περασμένο χρόνο είχαμε τα προβλήματα με τα ασφάλματα στο παράρτημα 7 Πού είναι όμως τώρα, γιατί τώρα πια δεν είναι αυτός ο κατάλογος στο παράρτημα 7, πού θα το βρω. Grazie. Passiamo adesso al punto presente il responsabile della Corte dei Conti Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να παραστώ εδώ σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων για το έγγραφό μας που αφορά, όπως είπατε και εσείς, ε, την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελληνικού Συνεδρίου 2 Κάστος 2010 από τα σημαντικά του καθιστών στήριξη για μελέτη σχεδιασμού και κατασκευή νέων υποδομών δυνάμει του έκτου προγράμματο πλαισίου έρευνα. Αυτά είναι τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτικής για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής διάστασης. Κατά την περίοδο 2002-2006 και υπό το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο η Ένωση πλήρωσε 140 εκατομμύρια σε ερευνητικά προγράμματα. Όπως λέει στο έγγραφό του και ο κύριος Κυλακάκης, πρέπει να δούμε αν τα δύο αυτά προγράμματα πέτυχαν το στόχο τους για την υψηλότερη δυνατή ιότητα με βάση μάλιστα τις ανάγκες που εξέφρασε η ερευνητική κοινότης. Θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα της εκθεσής μας θα είναι χρήσιμα για τους για όσους παίρνουν αποφάσεις και για να δημιουργήσουν τις κατάλληλες υποδομές. Επίσης εξετάσαμε το σημαντικό θέμα της προώθησης από την Κομισιόν της χρήσης συμπληρωματικής χρηματοδότησης για την έρευνα. Τα δύο αυτά προγράμματα ελέγχθηκαν με τα γνωστά κριτήρια, αλλά όπως είπε και ο συντάκτης της δεν, δεν ε, δεν υπάρχει σαφής αναφορά της ευρωπαϊκής υπεραξίας ή διάστασης και αυτό καθιστά την αξιολόγηση πιο δύσκολη. Οι ελεγκτές χρησιμοποίησαν τις μεθόδους που ξέρουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν έπαιξαν και αυτές το ρολάκο τους. σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες έγιναν επιτόπιοι έλεγχοι. Οι συντονιστές ερωτήθηκαν, ανακρίθηκαν για τα αποτελέσματα των ερευνών τους και τα κράτη-μέλη παίζουν κύριο ρόλο στην εφαρμογή τέτοιων νέων υποδομών και με ερευνητικά ιδρύματα μαζί που παίζουν ένα ρόλο στην Ένωση. Εμείς θεωρούμε ότι αυτά τα είχε δει με θετικό βλέμμα το συνέδριο και είχε ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ ερευνητών και ερευνητριών. και έτσι νομίζω ότι στηρίξαμε επικοδομητικά τα ερευνητικά προγράμματα που υπήρχαν. Όσο για τα νέα προγράμματα υποδομών, δεν ήταν προφανές, προφανής η χρησιμότητά τους. Η χρηματοδότηση κατά 10% για να χρησιμοποιηθεί ως καταλήτης δεν αποδείχθηκε. Τέλος, το συνέδριο κατέληξε ότι η χρησιμοποίηση διαφορετικών πόρων και πηγών πόρων δεν εφαρμόστηκε από την Κομισιόν. Γι' αυτό στις συστάσεις του το συνέδριο θεωρεί ότι η Κομισιόν πρέπει να δει κατά πόσον σε τέτοια προγράμματα δεν πρέπει να χρηματοδοτούν Τούνται αυτά από τον υπάρχοντα προϋπολογισμό της έρευνας. Δεδομένου βέβαια ότι θα γίνεται και μία εκ των υστέρων αξιολόγηση. Ως προς τη χρήση πρόσθετων πηγών πόρων, η Κομισιόν θα έπρεπε να δει τι μπορεί να επιτευχθεί από την επαναχρησιμοποίηση θέσεων του προϋπολογισμού εφόσον θεωρεί ότι θα είναι χρήσιμο. Με χαρά σημειώνω ότι το έγγραφο του κυρίου Σκυλακάκου τονίζει ότι πρέπει η Κομισιόν να αποδείξει ότι έχει κάνει την καλύτερη δυνατή χρήση των κονδυλίων της. Επίσης χαίρομαι διότι ο εισηγητής ο ίδιος κύριος Κυλακάκης υποστηρίζει την ιδέα ότι τα ωφέλη από τη χρήση συμπληρωματικής χρηματοδότησης πρέπει να γίνουν σαφέστερα και να θεωρείται η χρήση αυτή ως ζωτικός παράγων για την υποδομή της έρευνας. Σας ευχαριστώ.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 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι εξετάζουμε εδώ το θέμα της διαχείρισης της έρευνας. Με την έρευνα έχουμε ένα πρόβλημα στην πολιτική, γιατί υπάρχει ασυμμετρία τη πληροφορία μεταξύ ημών που εκπροσωπούμε τους φορολογούμενους και εκείνους που εισπράττουν τα χρήματα αυτά και τα δαπανούν για την έρευνα. Βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση όταν πρέπει να κρίνουμε κατά πόσο τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν όπως έπρεπε ή όχι. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να ελέγχουμε και να εξετάζουμε πώς δαπανήθηκαν τα χρήματα πιο λεπτομερώς στην έρευνα παρά σε άλλους τομείς όπου υπάρχει ανταγωνισμός. Για την έκθεση αυτή λέμε ότι το ενεργητικό συνέδριο εξέτασε διαφορετικά τις μελέτης ε, προετοιμασίας όπου τα πράγματα ε, ήταν αρκετά καλά και τις νέες υποδομές όπου λέει ότι δεν υπήρχε καμία προστιθέμενη αξία. Υπήρχε ζήτηση μεταξύ της Κομισιόν και του Ελεκτικού Συνεδρίου το τι σημαίνει προστιθέμενη αξία. Και η Κομισιόν είπε προστιθέμενη αξία σημαίνει να αυξηθεί η ευρωπαϊκή διάσταση. Όταν ακούω τέτοια πράγματα είμαι πολύ φυλακτικός τι θα πει ευρωπαϊκή διάσταση. Θα ήθελα από λοιπόν να ζητήσω από την Κομισιόν να μας πει λεπτομερώς πώς καταμετρά την ευρωπαϊκή διάσταση. Γιατί πολλά θα πανούμε για την ενδυνάμωση αυτή της ευρωπαϊκής διάστασης. για ε, μελέτες για την ε, τον συνδυασμό έκανε πολλές ε, συζητήσεις, επαφές κλπ. λοιπά. παρ' όλα αυτά, εγώ δεν βλέπω να αναφέρεται εδώ τίποτα για έναν έλεγχο αποτελεσματικότητας. Δηλαδή πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα αυτά όχι κατά πόσον μόνο δαπανήθηκαν προς τη σωστή κατεύθυνση για το σχεδιασμό στην προηγουμένη περίπτωση, αλλά κατά πόσον υπήρχαν υπερβολικά υψηλά κονδύλια για κάποιες μελέτες. Δεν νομίζω ότι έγινε κάτι τέτοιο, αλλά θα πρέπει νομίζω στα προγράμματα αυτά ε, να δούμε πού μπορεί να υπάρχουν σπατάλες, γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Έχουμε ίσως εσφαλμένους αιτιολογήσεις, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πιο λεπτομερείς στους ελέγχους εδώ, περισσότερο από ότι για άλλα είδη δαπανών. Ευχαριστώ πολύ. είναι